Έρχομαι τώρα στην ημερήσια διάταξη να σας παρουσιάσω. Την έχετε ε, στα χέρια σας ε, και να δούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Διαδικαστικό. Ναι, ο κύριος Λάχης. Καλά ε, κάνετε που μας συγχαίρετε που είμαστε παρόντες και ωραίο, αλλά ήταν επίπονο και καθήκον μας είναι. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Μόνο για την επόμενη φορά θα ήθελα να προτείνω κάτι το καθήκον αυτό να μας το διευκολύνετε λίγο ενημερώνοντάς μας ε, εγκαίρως, να απαντάτε και στα email μας και να ξέρουμε τι τρέχει και τι συμβαίνει. Και μπορεί να είναι παρόντες και όσοι απουσιάζουν σήμερα σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, οφείλω να πω ότι δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά την παρατήρησή σας πολύ καλά δράσατε και αντιδράσατε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι προτείνετε. Καλά, ας το αφήσουμε αυτό προς το παρόν και να ασχοληθούμε με την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να πω για τον συνάδελφο ότι ναι, υπάρχουν προβλήματα είναι οι νέε μεταφορές, Ανόητοι δεν είμαστε, αλλά γιατί έπρεπε να περιμένουμε σήμερα για να το διαπιστώσουμε αυτό. Αφού υπάρχουν τα προβλήματα, ναι, έστω κάποιοι ε, δεν έχουν έρθει, αλλά εμεί είμαστε εδώ. Έχει κοστίσει εκατομμύρια Βρετανικών λιρών όλη αυτή η υπόθεση στον ε, πολίτη της Ευρώπης και εσείς αποφασίσετε να καταργήσετε τις ψηφοφορίες. Ναι, ξέρουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες, αλλά εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι είμαστε κοινοβούλιο. Το μόνο που μας λέτε λοιπόν είναι ότι μπορούμε να έρθουμε να μιλάμε και μετά να ψηφίζουμε, να μην λαμβάνουμε αποφάσεις. Ο φορολογούμενος τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο αισθάνεται αποτροπιασμό όταν ακούει τέτοια πράγματα όταν έχουμε προβλήματα οικονομικά, όταν περιορίζουμε τις, την παροχή των, το, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όταν έχουμε εκλογές και τόσα προβλήματα, μας λέτε ότι με τόσα έξοδα που έχει προκαλέσει αυτή η σύνοδος θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Λέει ο Πρόεδρος. Όλες οι παρατηρήσεις είναι για μένα εξίσου σημαντικέ, λαμβάνω εξίσου υπόψη. Πλην όμω έχουν συμφωνήσει για τι προτάσει που θα σα παρουσιάσω τώρα για τι τροποποιήσει στην ημερήσια διάταξη. Έχουν συμφωνήσει όλε τι πολιτικέ ομάδε και μου επιτρέπετε να περάσω τώρα στην ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σοφή απόφαση να αναβάλουμε τις ψηφοφορίες γιατί μπορεί να υπάρχει απαρτία αλλά δεν υπάρχει γεωγραφική εκπροσώπηση σωστή. Την υπόλοιπη ημερήσια διάταξη όμως ε, ε, τη βλέπουμε ε, να περιορίζεται. Παρακαλώ να τη συμπιέσετε, να τελειώσουμε την Τετάρτη το μεσημέρι και όχι την Τετάρτη το βράδυ, να μην υποχρεωθούμε να μείνουμε και την Πέμπτη για να γυρίσουμε σπίτι μας. Κυρίε και κύριοι, θα σας παρακαλέσω να κοιτάξουμε τώρα την ημερήσια διάταξη. Σημείο προς σημείο. Και δίνω το λόγο μετά στους βουλευτές για τις παρατηρήσεις τους. Δευτέρα. Δεν υπάρχουν αλλαγέ. Όπως έχετε την ημερήσια διάταξη παραμένει. Γιατί την Τρίτη. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη δουλειά μας. Επιτρέψτε μου να προχωρήσω και να εξετάσουμε την ημερήσια διάταξη. Mr. please. Ναι, να σας πω όμως το εξής, χωρίς να το θέλουμε. Ενώ μεταφέρετε αυτή την ψηφοφορία για τις 6 του μηνός, ε, συμπίπτουν οι ψηφοφορίες που δεν γίνονται αυτήν την εβδομάδα την ημέρα των εθνικών εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μπορείτε να τις κάνετε τουλάχιστον στις 5 του μηνός Τετάρτη και όχι 5, η στις 6 του μηνός Μαΐου. Για να μπορούν να είναι και οι εδώ. Και οι Βρετανοί εδώ. Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι. Να σας πω. Θα επανέλθουμε στην υπόθεση αυτή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Επιτρέψτε μου να προχωρήσω και όταν τελειώσουμε αυτό το θέμα θα το ξαναδούμε με τη σειρά. Προς το παρόν δεν χρειάζεται να δούμε τις συγκεκριμένες ημέρες. 5 ή 6 Μαΐου θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Επιτρέψτε όμως να περάσω στην ημέρη ένταξη και δεν θέλω άλλο διαδικαστικό παρακαλώ. Και τώρα. Είπαμε τη Δευτέρα, έχετε την ημέρη δέταξη, δεν αλλάζει τίποτα. Για τη Δευτέρα δεν υπάρχουν τροποποιήσεις. Τρίτη. Αρχίζουμε στις 9 το πρωί με